Συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε, θα αρχίσουμε όπου να είναι. Ετοιμάστε τις κάρτες σας. Θα σας διαβάσω την ψηφοφορία τη σειρά τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικού ιατρικούς σκοπούς. Η συνάδελφος Ρης. Έπειτα θα ψηφίσουμε για την συνέχεια πρέπει να δοθεί στην εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και στον έλεγχο των κρατών μελών επί της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, τη δική μου έκθεση δηλαδή. Να το επαναλάβω. Όχι. Έπειτα, κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001-20 ε, Γκλένις μετά Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη, μια βιοοικονομία για την Ευρώπη, έκθεση του κ. Μπαρτολότσι και το κοινοτικό σύστημα καταχώρησης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών. Τη γνωμοδότηση της κυρίας Γιόρνταν. Είστε όλοι εδώ, ελπίζω. Μπορούμε να αρχίσουμε λοιπόν. Έκθεση ΡΙΣ. ψηφίζουμε συνολικά 1, 3, 4, 5 και 2 τις τροπολογίες αυτές υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οριστική ψηφοφορία ηλεκτρονικά όπως πάντα, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 32 ναι, κανένα όχι, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Ρης. Περνάμε στην επόμενη έκθεση. Τη δική μου έκθεση. Τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρο υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρο, υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, συνολική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση. Ψηφίσατε, πέρας ψηφοφορίας. 36 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σας. Προχωράμε τώρα το μεγάλο χοντρό βιβλιαράκι, έκθεση Wilmot. Ξεκινάμε αμέσω. 181. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές δεκτή. 182 και 186 μαζί. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. πέντε υπέρ, κατά. Αποχές, δεν είναι σαφές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 19 υπέρ 22 κατά απορρίπτεται. Δεν λειτουργεί το μαράφετ σας. Αλλάξτε θέση αν θέλετε. 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 184 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο παρακαλώ 184 άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 185 υπέρ Κατά. Αποχές δεκτή. 26 ΙΜΚΟ. Εκπίπτει. Όχι, όχι, πρέπει να το ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 187. Εκπίπτει. Την 188 υπέρ και 189 κατά. Αποχές απορρίπτονται. Απορρίπτονται. 188-189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 188-189. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Έγκρινεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. 193 υπέρ και ήμικο 28 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Θέλετε έλεγχο. 196 έλεγχος. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται όπως είπαμε. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 198 εν μέρη. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος, βεβαίως. 198, ναι, ναι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Δεχτεί. Ήμκο 29. Εκπίπτει. 199. Υπέρ. Αυτό είναι για αργότερα. Κατά. Απορρίφτεται. 200 εκπίπτει. υπέρ δεκτή 201 κατά αποχές δεν είναι σαφές 201 ελέγχουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας δεκτή 202, 204 και 30 που είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, δεκτή. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συγγνώμη. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Διακόσια έντεκα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 212 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.18 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.17 υπέρ. Έχω... Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Έλεγχος για 217. Ψηφίσατε όλοι. Όλες. Πέρας. Απορρίπτεται πράγματι. 2.19. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.20 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.21 2.22 συγγνώμη. Απορρίπτεται. Ήμκο 33 υπέρ. Κατά. Δέκα συνάδελφοι μονάχα έχουν ψηφίσει. Επαναλαμβάνουμε. ΥΜΚΟ 33 υπέρ. Κατά. Αποχές δεχτεί. Ήτρε 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.24 υπέρ. Κατά. Αποχές δεχτεί. 2.23 ήταν αυτή. Ηλεκτρονικά την ελέγχουμε. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. 34 εμικό. 2.24 και 25 πρέπει να ψηφίσουμε που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 2.26 και 1-15 ταυτόσιμες πάλι υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι, πέρας. Δεκτές. 2.27 και ΙΜΚΟ 35 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 2.28 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρικός έλεγχος στη 228. Ψήσατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.30 και ήτρε 17 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεκτές. 2.31 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.32 και ΙΜΚΟ 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Έλεγχος. 2.32 και ΙΜΚΟ 36 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται. Η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Οι σοσιαλιστές έχουν ένα που περισσεύει στην ψηφοφορία. Ένας ψηφίζει παραπάνω από τον αριθμό τους. Πρέπει να ξαναεπαναλάβουμε. Ψηφίσατε 36, ΙΜΚΟ και 223. 232 μάλλον. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Σαφώς εγκρίνονται. 2.34 και ΙΜΚΟ 37 σε τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά. Πολύ λίγοι συμμετέχουν υπέρ της 2.34 και της ΙΜΚΟ 37. Σηκώστε ψηλά τα χέρια παρακαλώ. Πολύ καλά. Κατά. Ωραία. Εγκρίνεται σαφώς. Δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά αποχές δεκτή, δεκτές. Έλεγχος στο δεύτερο τμήμα της ΣΥΜΚΟ 37 και της 234. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ψηφοφορίες. Εγκρίθηκαν. 20, 235 και ΙΤΡΕ 18. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 2.36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.37 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.38 δεν πρέπει να την ψηφίσουμε. Πάμε ή 19 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.39 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 12α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 20 το αντίστοιχο σημείο, το αντίστοιχο κομμάτι, πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2.46 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2.47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.51 υπέρ, κατά Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασ... Ε, παγιοποιημένη τροπολογία 3. Η Μαργαρίτα θέλει να κάνει μια προφορική τροποποίηση εδώ. Θα ήθελα να προτείνω μια προφορική τροπολογία στην ε, παγιοποιημένη τροπολογία 3 στο τέλος της πρώτης παραγράφου εκεί που θα λέγαμε βάση της δήλωσης του Διεθνούς Οργανισμού, Ιατρικού Οργανισμού στο Ελσίνκι η ίδια προσθήκη θα πρέπει να πάει στο τμήμα 2, στο εδρεωμένο τμήμα 2, παγιοποιημένο τμήμα 2. Όσοι εισηγήτρια το δέχομαι, λέει η κυρία Βίλμοντ. Ωραία. Με την τροποποίηση αυτή ψηφίζουμε την ε, παγιοποιημένη τροπολογιατρία υπέρ, κατά, απόχες με μεγάλη πλειοψηφία. 2.55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.56 και ΙΜΚΟ 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 2.57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πηδάμε στη διευθέτηση. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πετρεωμένη 25 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 272 και ΙΜΚΟ 41 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2,75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. Ήτρε ε, 21 υπέρ. Κατά. Ναι. Σελίδα 14 στο δικό μου κείμενο. Από την αγαπημένη μας, την προσφυλή μας Ήτρε, τροπολογία 21, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Εδρεωμένη 26, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 278 υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. 283 υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. 286 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 του εισηγητή υπέρ. Τι εισηγητές μου. Κατά. Αποχές δεκτή. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Το δεύτερο θύμα της 289 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 295 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρουμε ηλεκτρονικός έλεγχος 295 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στη 2.93 και την 3.24. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 2.97 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 2.98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές τρίτη. 2.99 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Έλεγχος για τη 299 αυτή ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Δεκτή. 300. Και η 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 301 και 245 45 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Στη συνέχεια το υπόλοιπο 302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Καλά, να ελέγξουμε. 27 και 303. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Σαφώς γίνεται δεκτή. 304. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 307 πρώτο τμήμα και 246 46 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 306 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 307 δεύτερο τμήμα, 26 δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συνεχίζουμε και πηγαίνουμε με την παγιοποιημένη 27 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 247 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παγιοποιημένη 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παγιοποιημένη 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 49 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για τη 49. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τρία δεκαεννιά υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 26 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήτρα 23 υπέρ. Όχι. Πρέπει να ψηφίσουμε την e 23, όχι την e 26. E23 23 λοιπόν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 εκπίπτει. 323 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 326 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Παγιοποιημένη 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 327. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμπκο 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3, 29 και 55 ΙΜΚΟ, ψηφιπέρ, κατά, αποχές δεν γίνεται δεκτή. Έλεγχος, έλεγχος 329 και ΙΜΚΟ 55. Ηλεκτρονικός έλεγχος, ψηφίσατε όλοι, πέρας πληροφορίας. εγκρίνονται. 3.30 υπέρ. Κατά. Απόχες. απολύπτεται. 3.31 ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. 3.32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.33 και 3.34 καθώς και η 3.27 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Λίμπε 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29. της συγκέντριας υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παγιοποιημένη 32 υπέρ κατά δεκτή. 3.42 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3.43 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3.45 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήμκο 58 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3.46 και ήμκο 60 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. 346 και ημικο 60. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνω την ψηφοφορία. Εγκριθήκανε. 347, 348 από κοινού ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 3.50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.53 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3.55 και υπέρ 30 από κοινού υπέρ, ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτονται. 3.54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 3.57 και ΙΜΚΟ 62 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτές 3.58 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ήτρε 31 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 3.59 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3.60 και ΙΜΚΟ 61 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεκτές. 3.61 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3.62 και ΙΜΚΟ 63 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 364 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 363 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 365 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 366 και ΙΜΚΟ 65 υπέρ. Κατά απόχες δεκτές. Παγιοποιημένη 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Κάνουμε ένα μικρό άλμα. Τρία 81, σελίδα 27 για μένα. Τη βρήκατε? Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έχουμε κάνει το πρώτο τρίτο, λέω. ο Θέλουμε καμιά ώρα ακόμα. Κουράγιο. 384 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 382 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 34 υπέρ. Εκπίπτει. Εκπίπτει, ναι, συγγνώμη. Εκπίπτει 34. 387 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 388 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά για 388. Ψήφισατε όλοι. Κλείνω την ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 389 και η 33 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.90 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 3.91 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 35 και 34 ε, της Ήτρα. Όχι, όχι. Συγγνώμη. Μόνο 35. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται εκπίπτει ως εκ τούτου η 34. 392 καθώς και η 35 υπέρ κατά αποχές δεκτές 393 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3.94 και M71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.95 και ίτρε 36 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 3.95 και ίτρε 36 ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνονται. Συνεχίζουμε. Ήμκο 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 396 εκπίπτει Ήτρε 37. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήτρε 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προχωρούμε με την 400 υπέρ και η 340 κατά αποχές απορρίπτεται. Η 341 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 342 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 404 και 401 υπέρ κατά αποχές δεκτές 405 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 406 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 407, 408 και 73 ψήφι υπέρ κατά. Αποχές δεκτές. Παγιοποιημένη 5. Με προφορική τροποποίηση ακριβώς την ίδια που είχαμε στην παγιοποιημένη τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 410 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πάγιο ποιημένη 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 411. 414 συγγνώμη. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 416 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 418 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 419 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παγιοποιημένη 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 421 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 422 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 423 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 424 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Παγιοποιημένη 35 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 425 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Δεν είναι σίγουρο, εντάξει έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος 425. Έχετε ψηφίσει όλοι. πέρα Πέρας προφορίας. Δεκτή. 428. Υπέρ. Κατά. Αποχέ Απορρίπτεται. 427. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παγιοποιημένη 36 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 4.30 δεύτερο τμήμα και η 4.29 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 4.31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε,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 39 ηλεκτρονικό έλεγχο Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι πέρα ψηφοφορία. Δεκτή. 346 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 4, 432 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 41 υπέρ. Κατά αποχές. 4.42 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 4.45 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 47 ε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, 42 υπέρ κατά άποχες γίνεται δεκτή. Και ερχόμαστε 494 και ΙΜΚΟ 76 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 450 και ΙΜΚΟ 77. 455 συγγνώμη και 97, 79 ΙΜΚΟ από κοινού. Κατά. Δεκτές. 43 υπέρ Συγγνώμη, πάω 4.45 ε, πάλι. Δεν την ψηφίσαμε. Κατά. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4.53 ίνκο 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος καλύτερα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Συνεχίζουμε. 4.54. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 456 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 440 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 48 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 457 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 458 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 459 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 460 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 47 ε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 470 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παγιοποιημένη 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη Λίμπε 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 474. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 4,75 ΙΜΚΟ 81 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4,78 καταπίπτει. Ψηφίζουμε Η 4,76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πίπτη 478. 477. Ένα μέρος της υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 479 και ΙΜΚΟ 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 480 ΙΜΚΟ 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 482 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 483. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Όχι, συνεχίζουμε με 484. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 485 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 484 και 485 πέρας ψηφοφορίας. Εισηγήτρια, νομίζω πως έχουμε λάθος νούμερο. Ποιο νούμερο ήταν, διότι στα αγγλικά μας είπαν κάτι άλλο, λέει η εισηγήτρια. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ψηφίσαμε την 485. Μήπως ήμουν γρήγορο, 485. Να την επαναλάβουμε καλύτερα. Ψηφίζουμε για την 485, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται, όπως και πριν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο πιο αργά. 486 και 501 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 487 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 491. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την τροπολογία 492 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος 482. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 493 και ΙΜΚΟ 85 με μια προφορική τροπολογία των πρασίνων. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 494. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Λίμπε 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 496. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 497. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 499. Ψηφοφορία σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κοιτάξουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 499. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 500. Και ΙΝΚΟ 84 καταπίπτουν 502 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε συμβιβαστική 21, 22, 23 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. ημίχρονο, 45 λεπτά, αρχίζω και βαριέμαι. Συμβαστική 19, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 520, απορρίπτεται. 518 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 518. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 521. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 522. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 523 και ΙΝΚΟ 94 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 524 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 526 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Χωρίς να ψηφίσει ο κύριος Ζέμπερ. Ο κ. Σνέλχαρτ, ηλεκτρονικός έλεγχος 526. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 525 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα λοιπόν Πάμε στην σελίδα 50, τροπολογία 53. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 544 καταπίπτει, 543 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμκο 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5.45 και ΙΝΚΟ 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 5.47. ΙΝΚΟ 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5.48. Υπέρ. Κατά. Παρακαλώ. Πιστεύω πως υπάρχει κάποιο λάθος. Ποια ψηφίζουμε ακριβώς. Υπήρξε... ένα πρόβλημα διερμηνία, ε, ενώ νομίζαμε ότι ψηφίζαμε για το 546 ενώ ψηφίζαμε για την 547. Θα ήθελα να ξαναψηφίσουμε. Βλέπω πως δεν πρέπει να ψηφίσουμε την 546, αλλά την 547 και ΙΝΚΟ 98. Αν θέλετε το κοιτάζουμε ηλεκτρονικά. Ηρεμήστε, ξέρω ότι έχετε ένα το αλλά ηρεμήστε. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. 547, ΙΝΚΟ 98. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 548 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπα 6. Χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτό. Ήτρε 52 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 5.50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5.51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος 551. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 552 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 553 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 554 και 555 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 556 υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 557, 558 και ΙΜΚΟ 99 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 559 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 560 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 561. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 54 καταπίπτει. 564 και ΙΜΚΟ 102 τώρα. Λοιπόν, Μάλιστα. 564 και 102 είχα δει και από την αρχή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 565. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 566. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 572. Υπέρ. 570. Με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 572 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερις ώρα περιμένουμε τον καφέ. Ίνκο 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 8 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 574 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 575 και ημικό 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 576 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 577 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 579 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 582. Υπέρ. 582. Επαναλαμβάνω. Και στα αγγλικά. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 582. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 583. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 586. Πρόσθετο τμήμα. Υπέρ. Κατά. 586. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 587. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 588. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 589. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57. Υπέρ κατά, εγκρίνεται. 58, 590 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Ίνκο 107, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μάλιστα ηλεκτρονικός έλεγχος, όταν ο πρόεδρος έχει ερωτηματικά, κοιτάζουμε και ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 591. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ίνκο 108. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 594. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5.95. Υπέρ. 5.95. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5.96. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59. Με μια προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος 59 με την προφορική τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Άρα, τώρα ψηφίζουμε την 59 χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Και αυτή απορρίπτεται. 597 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 598 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 599 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 601 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 605 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 606 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 608 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 607. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 609. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 610. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 611. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6-12. Υπέρ. κατα αποχης Αποχές. Απορρίπτεται. 6-13 και ΙΜΚΟ 110. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 6-14 και ΙΤΡΕ 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 6-15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές 617. υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ποια. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 61. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 6-17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6-18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6-19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6-20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6.21-6.22 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβιβαστική 38, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παγιοποιημένη 39, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6.35, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος 635. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε 642. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113. Ήμκο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6.43. Ίνκο 113. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 6.43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6.44 και 6.45 μαζί, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ήτρε 55, υπέρ. Όχι, Ήτρε 55 καταπίπτει. 6.46, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται αλλά θα κοιτάξουμε ηλεκτρονικά την 646. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 647 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 649 και ήτρα 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 650 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνονται. Λίμπε 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 651, 655, υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 652, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 653, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 654 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 57 υπέρ. Κατά. Αποχές επορρίπτεται. Ήτρε 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παγιοποιημένη 40 στην σελίδα 64. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Παγιοποιημένη τροπολογία 40. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε 661, 662, 663, 666, όλες μαζί, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 65. Και η 359 μαζί. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Εγκρίνονται. 1664 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πέρας πληροφορίας. Απορρίπτεται. Μάλιστα, αρχίζει από μόνη της ηλεκτρονική ψηφοφορία, βλέπω. Συνεχίζουμε, ήτρε 60, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 665 και ίνκο 114, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνονται. 667, υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπα 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 669. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμικο 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 670. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος στην 670. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. 671. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 672. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπα 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την 446, το ανάλογο κομμάτι, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. «673. Υπέρ κατά, αποχέ εγκρίνεται. 674, 675 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 677 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 678 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ή ηλεκτρονικός έλεγχος για την 678. Πέρας. Εγκρίνεται. 6,79, 6,80 μαζί υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτονται. 681 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 682 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1 τμήμα της ΙΝΚΟ 116 υπέρ, κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ίνκο 116, δεύτερο μέρος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 684. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 685. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 686. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 687. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 688. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 689. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 6.90 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6.91 και η 3.63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ήμικο 117 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6.92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ίνκο 118 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 695 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 696 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 697 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 699 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 700 υπέρ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ίνκο 120. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 701. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 702. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπε 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 703. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 704. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 705. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 706. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 707. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 708. Το υπόλοιπο του κειμένου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 709. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 710 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72 και 711 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Νόμιζα πως είχε εγκριθεί. Ας το κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 7-12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7-13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7-13 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 7-14. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7-15. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7-16. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 7-17. Το υπόλοιπο του κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 πίπτη 73 υπέρ. Κατά. Αποχής. εγκρίνεται. 7, 74. Θέλω καφέ, λέει ο πρόεδρος. <laughs> Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ηλεκτρονικός έλεγχος στην 74. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 7-19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπε 15, λίμπε 16 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 7-20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 721 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 722 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 723 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 724 και 121 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 725 υπέρ Ηλεκτρονικός έλεγχος 724 και 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 725 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 726 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπα 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 727. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 728. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 729. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 730 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 123 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ήμκο 124 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 125 γιώτα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ή τρένα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 και ενικό ένα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. 84 ηλεκτρονικός έλεγχος. Βεβαίως. Πέρας. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 87. Ψηφίσατε. Πέρας. Πράγματι απορρίπτεται. 88. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τρία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ήτρε Τρία. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 97 δεν θα τη ψηφίσουμε. 98 πάμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απο... Εγκρίνεται. Ήτρε 5 καταπίπτει. Ήμικο 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 και η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105 και 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε την 112 και προχωράμε στην 114 να κοιτάξουμε. 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Όχι. Όντω 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήμκο 8 καταπίπτει και η τρέπτα. Επιτέλους ήρθε ο καφές. 115 και ήμκο 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 και η τρέξη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ήμκο 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παγιοποιημένη 6. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 13, ήμκο, υπέρ, καταπίπτει, 13, Ήμκο 15 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παγιοποιημένη 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχο καλύτερα για την 41. Ψηφίσατε όλοι. Παγιοποιημένη 41. Επαναλαμβάνω. Πέρας. Εγκρίνεται. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 132. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 134. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 20 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμικο 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1.44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 145. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκα... Απορρίπτεται. 146 και ήμικο 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 147. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 148 και 149 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 152 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 153 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 154 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 156 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 158. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. 159 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 160 δεν θα την ψηφίσουμε. Ψηφίσουμε την 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 164 και 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 167. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 168. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ήμικο 24. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 170. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 171. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λιμπένα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 173, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 174, υπέρ, το υπόλοιπο του κειμένου, κατά, δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος 174. Πέρας. Εγκρίνεται. 1,75. 1,76. Ίνκο 25. Όλες μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 1,77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος 177 και η 13. Πέρας. Απορρίπτεται. 178 και 179 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ουφ, λέει ο πρόεδρος. Οριστική ψηφοφορία. Η ηλεκτρονικά όπως πάντα άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 65 υπέρ, καμία ψήφος κατά. Πάμε τώρα μισό λεπτό. Δεύτερη ψηφοφορία, δεν τελειώσαμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 64 ψήφοι υπέρ. Και τώρα σας ερωτώ. Θα ήθελε η συγκήτρια να λάβει διαπραγματευτική εντολή στην πρώτη ανάγνωση. Γκλένης, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Να πω καταρχήν ευχαριστώ σε όλους τους τις συγητές για το θαυμάσιο έργο τους και τη συνεργασία τους. Ήταν μια μεγάλη χαρά να συνεργαστώ με όλους τους. Παρά το γεγονό ότι ήταν τεράστιο ο αριθμό των ε, τροπολογιών και πάρα πολλά προβλήματα, καταφέραμε να πετύχουμε μια ευρεία συμφωνία στα, σε όλα τα θέματα και προχωρήσαμε πάρα πολύ για τα θέματα Επιτροπής Δεοντολογίας και διαφάνεια σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο γιατί ο χρόνος προχωράει και τελειώνει ο χρόνος για τη δίκτυα αυτή του Κοινοβουλίου και είναι απαραίτητο να υπάρξει αυτή η νομοθεσία το ταχύτερο δυνατό. Υπάρχουν κάποιε ανησυχίε, το ξέρω, και είμαι ανοιχτή για να ακούσω τι απόψει αυτέ, αλλά όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι βιομηχανικοί κλάδοι, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, τα λόμπι, οι ακαδημαϊκοί, οι ερευνητές, όλοι θα ενοχληθούν και θα απογοητευτούν αν καθυστερήσει η πολιτική διαδικασία. Δεν πρέπει να την ανατρέψουμε λοιπόν. Ζητώ από όλους να υποστηρίξουν αυτή η διαπραγματευτική εντολή. Μπορούμε να ψηφίσουμε χωρίς να διακόψουμε λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία για την διαπραγματευτική εντολή. η, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 62 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Αγαπητή κυρία Βίλμοτ, σας ζηλεύω. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι με πνεύμα ευθύνης έχουν αντιμετωπίσει αυτή την εκθένη και διευκόλυναν το έργο μας και φυσικά και την ε, γραμματεία θέλω να ευχαριστήσω που προετοίμασε τόσο καλά τα, τα έγγραφα αυτά για να μπορέσουμε να κάνουμε πληροφορία. Συγχαρητήρια Κλένη. Συνεχίζουμε τώρα. Με την βιοοικονομία για την Ευρώπη, ο κύριος Μπαρτολότσι είναι ο εισηγητής στην έκθεση αυτή και συνεχίζουμε. Ε, τροπολογία της ΕΜΠΛ, της ε, απασχόλησης υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για 17 ψηφίσατε όλοι Πέρασε. απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η τρένα, υπέρ πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έμπλ 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 25. 25. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 29. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 32 τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 33 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 32 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. 31 ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικό έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 36 υπέρ. Έλεγχος για την 35. Μάλιστα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ήτρε 8. Δεύτερη φράση. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 30 συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ελεκτρονικό έλεγχος για 44 αρχή ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, κλείνω την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 47 υπέρ και ρεύγει 10. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ρέγγι 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έμπλ 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έμπλ 14 εκπίπτει. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για τι 48 ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 48 εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά. απόχέ δεκτή. Έμπλ 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέες απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχέες απορρίπτεται. 52. Υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές 52 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή έμπλε νέα, υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 12 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έμπλ 15 πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έμπλ 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 67. Υπέρ. Έλεγχος ήτρε 12, ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 13 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71ο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές δεκτό Ρέγγι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήτρε, 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 17, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές έλεγχος για το πρώτο τμήμα της Ήτρε 17, ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις πληροφορία Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Εμπλοκτό, υπέρ Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά. Εμπλοκτό. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Στο τσάκ απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πάμε στην 75 υπέρ. Κατά. Αποχές δεχτή. 10 την ψηφίσμου. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ρέγγι 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ρέγγι 7 υπέρ, έλεγχο στην ρέγγι 14, άρχεται, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας, απέριπτη. Ρέγγι 7 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Και εδώ έλεγχος, ρέγγι 7. Ψήφισατε όλοι, Πέρας. Είναι σαφές ότι απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά για την 82. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνω την ψηφοφορία. Α, απέριπτε. Έμπλη 10 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πάμε στην 88 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 87 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλεφτα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Παγιοποιημένη 6 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά, παγιοποιημένη τροπολογία 6. Ψήφισατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Παγιοποιημένη 7. Εκπίπτει. Ήτρε 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, δεν είναι σαφές. 95 ηλεκτρονικά. Ψήφισαμε όλοι. Πέρας. Ισοψηφία απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ήτρε 2 λέει ο πρόεδρος Συγγνώμη, 99, τροπολογία 99, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέκι 13, πρώτο τμήμα, υπέρ. Α, εκπίπτει, συγγνώμη, συγγνώμη, εκπίπτει. Όχι, όχι, πρέπει να την ψηφίσουμε. Σιγά σιγά, πιο σιγά. 99 απερίφθη, Επομένω, η Ρέκη 13 θα πρέπει να ψηφιστεί. Υπέρ. Κατά απόχες δεν είναι σαφές ηλεκτρονικά ρέγγι 13 ηλεκτρονικά ψήφισατε όλοι πέρας απορρίπτεται Ίσως Μπορούμε να διακόψουμε το πηγαδάκι και να συνεχίσουμε. Έμπλου 17 κατά αποχές δεκτή. Η τρενέα κατά αποχές δεκτή. 100 υπέρ. Κατά. Η τρενέα θέλετε έλεγχο ηλεκτρονικά. Εντάξει. Άρχισε η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τμήμα 1, παράγραφος 1, δεύε, δεύε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 6 της δεύε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την ε, παράγραφο 1, δεύε, ψηφίσατε όλοι, πέρας. Δεκτή. Παράγραφος 6 της δεύε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. δεκτή. 9 υπέρ. Την 7 την ελέγχουμε ηλεκτρονικά άρχιδη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. δβ 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεβε 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή δεβε 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεβε 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή δεβε 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ασαφές. Ηλεκτρονικά είναι 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ ελέγχουμε την 3 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται για μία ψήφο 4 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήτρε αιτιολογική σκέψη Β. Έλεγχος για την 6. Μάλιστα. Άρχεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήτρε Αιτιολογική σκέψη Β. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμπλε Κατά. σκέψη Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 10. Υπέρ κατά αποχές απολύπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απολύπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές απολύπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές 15 15 υπέρ. Κατά. Ε, εγκρίνεται. Ήτρε αιτιολογική σκέψη α υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήτρε αιτιολογική σκέψη σε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλ αιτιολογική σκέψη σε υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έμπλε τη λογική σκέψη δε... υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλε τη λογική σκέψη α, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλε τη λογική σκέψη ε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλε τη λογική σκέψη F, σίγμα τάφ, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. 54-0 με 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπορτολότσι. Είναι Morgen mit den Abstimmungen weiter um 10. Συνεχίζουμε αύριο στις 10 η ώρα τις ψηφοφορίες και θα έρθει τώρα η Επίτροπος, οπότε διακόπτουμε την ψηφοφορία. 10 η ώρα το πρωί θα συνεχίσουμε. So, ich bitte doch diejenigen, die... Μάλιστα. Συνάδελφοι, όσοι θέλουν να παρευρεθούν στη συζήτηση, να καθίσουν παρακαλώ. Και σιγά σιγά παρακαλώ να επικρατήσει η ησυχία. Ξέρω ότι ήταν τόσο ενδιαφέρον αυτό που κάναμε πιο πριν. Η ψηφοφορία ήταν δίωρη. Να καλωσορίσω τώρα την Επίτροπο Περιβάλλοντος, Κόνι Χέντεκαρτ, Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Πάρα πολλούς εφακέλους, ορισμένα θέματα τα συζητούμε δύο φορές, το backloading για παράδειγμα. Επίσης, την νομοθεσία σχετικά με τα φόρτικα και με τα ελαφρά οχήματα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα μέσα μιας οικονομικής κρίσης όπου το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος συγκρούεται με τα οικονομικά συμφέροντα. Δεν πιστεύω ότι όμως αυτό είναι κατά κακό. Μπορούμε να δούμε τους πόρους μας, και πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά, όχι μόνο το πετρέλαιο αλλά και το αέριο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον αλλά και το πορτοφόλι των καταναλωτών. Είμαι περίεργος να ακούσω τι έχει να πει λοιπόν η Επίτροπος. Φέτος η Διεθνής Διάσκεψη για το Περιβάλλον θα γίνει στην Βαρσοβία. Αν σας ενοχλούμε πείτε μας παρακαλώ. Το 2015 θα διεξαχθεί επίσης μια διάσκεψη στο Παρίσι και θέλουμε να δούμε πώς θα είναι η δική μας στρατηγική ως Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να επιτύχουμε μια παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. Ο Πατερλίζε, ο εισηγητής, είναι εδώ μαζί μας να σας πω ότι κάπως με ενόχλησε όταν διάβασα στην εφημερίδα ότι οι κατασκευαστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλαν μία επιστολή προς την Κίνα με την οποία ξεκαθάρισαν ότι η νομοθεσία εδώ πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ περίεργος να ακούσω τι έχει να πει η Επίτροπος για τα εκρεμή ζητήματα. Να καλωσορίσω λοιπόν την Επίτροπο και να της δώσω το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ματίας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Ματίας. Δεν νομίζω ότι είναι βαρετό, αλλά νομίζω πως πολλοί θα συμφωνούσαν σήμερα μαζί μου, αυτή την με την αίσθηση δηλαδή ότι κάποιες φορές το να μιλάμε για κλιματικές αλλαγές, το να περνάμε ε, ε, ε, νομοθεσία κατά των κλιματικών αλλαγών μπορεί κανείς να αισθάνεται πως αγωνίζεται πολύ σκληρά όμως κάποιες στιγμές συμβαίνουν πράγματα προχτές κάναμε μια συνεδρίαση στην Κομισιόν για τις συστάσεις αναχώρα και πραγματικά πολλές χώρες φέτος είχαν συγκεκριμένες συστάσεις να υποβάλουν ε, σε σχέση με το κλίμα, την ενέργεια, την ε, επάρκεια σε πόρους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι δηλαδή όντως κάτι κινείται. Φέτος πραγματικά πρέπει να αποδώσουν, διότι διαφορετικά θα έχουν να αντιμετωπίσουν τι επιπτώσει του χρόνου. Και επίσης την περασμένη εβδομάδα οι επικεφαλείς κρατών συζήτησαν την ενέργεια και υιοθέτησαν πολύ καλά συμπεράσματα του Συμβουλίου που λένε μάλιστα ότι το 2030 καλωσορίζουν τώρα το πράσινο βιβλίο, το ξεπέρασαν και εμείς σαν Κομισιόν πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να αποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις που μετά θα τις συζητήσουν τον επόμενο Μάρτιο. Σε μερικά μεγάλα θέματα λοιπόν προχωράνε τα πράγματα. Είναι καλό λοιπόν να πούμε δύο λόγια για ένα θέμα το οποίο ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πάντα σε αυτή την επιτροπή, είναι το backloading. Το έχουμε συζητήσει εκταμένα και στην ε, Ολομέλεια τον Απρίλιο και εγώ είχα επαφή με εκπροσώπους από πολιτικές ομάδες και μάλιστα υπάρχει ένα έγγραφο με στοιχεία. Ό,τι και αν πιστεύει κανείς για αυτό το θέμα, καλό είναι να γνωρίζει ακριβώς περί πρόκειται και να μιλήσουμε σωστά για τις αναλογίες. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθώ επίσης εδώ να πω ότι τα πρόσφατα στοιχεία από τις ε, συναλλαγές που έγιναν, ε, από τότε που κάναμε την πρότασή μας, η υπερβολική παροχή στο σύστημα δεν έχει μειωθεί, έχει αυξηθεί μάλιστα κατά 2 δισεκατομμύρια. Και πάλι αυτό το λέω για να έχουμε υπόψη μας τις αναλογίες. Καλωσορίζω λοιπόν την απόφαση των συντονιστών της ΕΝΒΗ να δουλέψουν για μια διορθωμένη ε, τροποποιημένη έκθεση που θα υποβληθεί στην Ολομέλεια και ότι θα, ε, που θα συζητηθεί τον Ιούνιο στην Επιτροπή για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να έχει μια άνετη πλειοψηφία και για τις τροπολογίες ε, φυσικά είμαι ανοιχτή να συζητήσουμε και νέες ιδέες που μπορεί να προταθούν εν ώψη της ε, ε, αναζήτησης συμβιβασμού. Νομίζω ότι όσο πιο γρήγορα συμφωνήσουμε τόσο καλύτερα για να μπορέσουμε να εστιάσουμε την προσοχή σε δομικά διαρθωτικά μέτρα και να σχεδιάσουμε πιο μακροπρόθεσμα την πολιτική μας. Φυσικά και προσβλέπω στα σχόλιά σας για την έκθεση περί κοινής αγοράς καθώς και τις διαρθωτικές αλλαγές που προτείνουμε εδώ. Ε, φαντάζομαι ότι αυτές θα τις αναμένουμε μετά από το καλοκαιρινές διακοπές και πάλι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ήταν ξεκάθαρα την περασμένη εβδομάδα εξφράστηκε η ισχυρή υποστήριξη σε μια καλά λειτουργούσα κοινή αγορά. Για το πλαίσιο πολιτικής μέχρι το 2030 ακτιμώ την προσπάθεια του Κοινοβουλίου να ε, αναπτύξει ένα πλαίσιο πολιτικής για τις εκπομπές και είναι σαφές ότι θα πρέπει να ορίσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα το μπλε βιβλίο για τις εκπομπές αερίων του, διοξίου, ε, αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030. Επίσης για τις ανανεώσιμες είναι σαφές ότι χρειάζονται νέοι στόχοι για τις ανανεώσιμες μέχρι το 2030 και εδώ επίσης πρέπει να προβληματιστούμε πώς μπορούν οι ανανεώσιμες, ε, η επάρκεια και ε, το διοξίδιο μπορούν να, να, να επηρεάζουν το ένα το άλλο, να συντονίσουμε τις πολυσχετικές πολιτικές. Δηλαδή αυτό το κάνουμε στην Κομισιόν και εδώ και ξε... γι' αυτό και ξεκινήσαμε και το πράσινο βιβλίο και είχαμε και με κάποιες προκαταρτικές σκέψεις από πλευρά των Ευρωπαίων ηγετών την περασμένη εβδομάδα. Τονίζω επίσης τη σημασία του να υπάρξει μια ενημερωμένη συζήτηση για αυτά τα θέματα στο Κοινοβούλιο και νομίζω ότι μετά τη συνεδρίαση των αρχηγών κρατών την περασμένη εβδομάδα δεν είναι το θέμα του αν θα έχουμε τέτοια πολιτική αλλά πώς θα είναι αυτή, ποιοι θα είναι οι στόχοι, ποια θα είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ τους και φυσικά ποιο θα είναι το επίπεδο ε, φιλοδοξίας. Ε, αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα. Περιμένω χρήσιμη ανταπόκριση από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα υπάρξει και μια διάσκεψη των ενδιαφερόμενων φορέων τον Ιούνιο και τα αποτελέσματα φυσικά θα συμπεριληφθούν και στην αξιολόγηση αντικτύπου για την προετοιμασία των πρωτοβουλειών μέχρι το τέλος του έτους. Δύο λόγια γιατί αναφέρατε και το ETS και την, την αεροναυτιλία. Ε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι εγκρίθηκε γρήγορα και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό γιατί μας βοήθησε πολύ. Νομίζω πως το Κοινοβούλιο δικαίως τόνισε πως Ε, το πάγωμα του χρόνου είναι μια περιορισμένη λύση χρονικά. Χρειάζεται να βρεθούν λύσεις ε, και μια πιο μόνιμη μάλιστα λύση του θέματος. Οι συνομοθέτες δήλωσαν ότι δύο συγκεκριμένοι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν μέσω της ΙΚΑΟ. Καταρχήν ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη μιας ε, ενός διπλού μέτρου μέτρησης της αγοράς και δεύτερον επιπτώσεις ε, στα, των μέτρων στη διεθνή αεροπλοεία με βάση, ε, μάλλον εφόσον εκκρεμεί η εφαρμογή του παγκοσμίου συστήματος. Η συμφωνία για τα μέτρα με βάση την αγορά θα πρέπει να διευκολύνει τις χώρες και τις περιφέρειες ώστε να προβούν σε, σε αποτελεσματικές δράσεις άμεσα. Ταυτόχρονα περιμένουμε από τους εταίρους μας και από τον κλάδο να συμφωνήσει ότι ένα παγκόσμιο σύστημα είναι η καταλληλότερη λύση. Η ΚΑΟ θα πρέπει να ξεπεράσει αυτή την ανάγκη, να το εξετάσει ως πακέτο, εξετάζοντας το βρέχεις πρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η Κομισιόν να προτείνει νομοθετική δράση ώστε να υπάρξει ένα επιτυχές και απλό αποτέλεσμα. Ε, βέβαια δεν χρειάζεται να πω, είναι αυτονόητο ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτός ο αγώνας. Πολλή δουλειά γίνεται αυτή τη στιγμή. Μπορώ να πω απλά ότι τα όσα κάνατε εσείς εδώ σε αυτήν την Επιτροπή που μας βοήθησαν και ξέρω πως υπάρχει και μια αντιπροσωπεία που πηγαίνει μεταξύ άλλων και στη ΣΥΠΑ ε, σύντομα και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν πως η νομοθετική μας συνέλευση έχει συγκεκριμένες απόψεις και σταθερές απόψεις. Να στραφώ τώρα σε κάποια άλλη πρόσφατη πρωτοβουλία. Πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δέχτηκαν την πρόταση της Κομισιόν να υποβάλουν τουλάχιστον το 20% μάλλον να αφιερώσουν σε δαπάνες σχετικές με το κλίμα το 20% του προπολογισμού για τα επόμενα 7 χρόνια. Και για μένα αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα, αλλά με το ότι δείχνει μια αλλαγή στην οτροπία και στη σκέψη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλοι αυτέ οι φιλοδοξίε θα αντικατοπτρίζονται σε σαφή στόχο, σε διαφανή σύνολα μέτρων, σε όλε τι σχετικέ πολιτικέ και προγράμματα. Αυτό είναι το CAP, το Horizon 2020, η πολιτική συνοχή, η διευκόλυνση Connecting Europe, ε, όλα αυτά τα, όλες αυτές τις κεντρικές πολιτικές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτή τη δέσμευση. Έπειτα υπάρχουν ε, ε, νομοθετικές προτάσεις στη διαδικασία συναπόφασης. Ο πρόεδρος ήδη ανέφερε την έναρξη του τριμερούς διαλόγου για κάποιες από αυτές πρέπει να βρεθούν πολιτικές λύσεις για να βρεθούν ε, συμφωνίες για την πρώτη ανάγνωση. Καταρχήν ε, τα super credits, μετά οι διαδικασίες ελέγχου των ε, οχημάτων και έπειτα τι θα γίνει μετά το 2020. Η Κομισιόν οφείλει να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο για να βρει αποδεκτή συμβιβαστική λύση μέσα στους επόμενους μήνες. Βιοκαύσιμα Τα βιοκαύσιμα είναι ένα περίπλοκο θέμα. Πρέπει να βρούμε τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούμε είναι πραγματικά βιώσιμα, ότι εκπέμπουν λιγοστά αέρια του θερμοκηπίου, περιβαλλοντικά είναι βιώσιμα και είναι και ανταγωνιστικά από άποψη κόστου. Γι' αυτό και θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα πιο βιώσιμα βιοκαύσιμα και η πρόταση που κάνουμε περιορίζοντα ε, τι πρώτε γενιά στα βιοκαύσιμα που βασίζονται σε, ε, ε, σε, σε παραδοσιακών ε, τροφίμων και να ενθαρρύνουμε τη δεύτερη γενεά. Βέβαια, θα συνεχίσει η Κομισιόν να εργάζεται για ένα φιλόδοξο αποτέλεσμα και φυσικά βασιζόμαστε τη δική σας υποστήριξη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, είναι τεχνικό, είναι δύσκολο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το φέρουμε σε αίσιο πέρας. Για το αέριο σχιστόλιθο έχουμε, ξέρουμε ότι μπορεί να σημάνει μήνυμο κόστος για το βιομηχανίες και αυτό θα είναι μια συμβολή που ευθυγραμμίζεται και με τον ε, οδικό χάρτη για χαμηλό διοξίδιο. Με την πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, επίσης με τη δέσμευση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στη μείωση των, φθοριούχων, των εκπομπών φθοριούχων αερίων έτσι ώστε τελικά να κρατήσουμε ηγετική θέση και να παρασύρουμε και άλλες χώρες στην πραγματική μείωση των εκπομπών φθοριούχων. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία πρώτης ανάγνωσης ε, το φθινόπερο πριν από την επόμενη συνάντηση των εταίρων για το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ. Τώρα, κλιματικές αλλαγές, ναι, με ανάβληση, αλλά και πιο επιθετική στρατηγική ε, δεν χρειάζεται να πούμε ότι υπάρχουν όρια στο πόσο περιοριστική μπορεί να είναι μια στρατηγική, ευρωπαϊκή στρατηγική προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, αλλά πρέπει πολύ περισσότερο να μοιραστούμε τις γνώσεις μας, να προετοιμάσουμε κατευθύνες γραμμές, ε, να μπορεί να είναι το θέμα των ασφαλιών, τα προβλήματα των παρακτήων περιοχών, ένα σωρό προβλήματα σε όλο αυτό το πακέτο μέσω κατευθυντήριων γραμμών θα τα αντιμετωπίσουμε και να πω και κάτι ακόμα, αυτή η πολύ ισχυρή σύσταση σε όλα τα κράτη-μέλη να φτιάξουν ένα συστημικό σχέδιο προσαρμογής πριν από το 2017. Αυτή τη στιγμή μόνο 15 κράτη-μέλη έχουν τέτοια προγράμματα. Προτάσεις για φέτος. Τώρα σύντομα, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, η Κομισιόν φυσικά είναι προσιλωμένη στην ανανεύρεση μιας παγκόσμιας λύσης για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την αυτιλία. Πρόσφατες συμφωνίες έχουν, είναι πολύ ενθαρρυντικές γιατί όλα τα μέτρα της αγοράς ε, συμπεριλαμβάνουν την παρακολούθηση, την ε, αναφορά αλλά και την επαλήθευση αυτών των εκπομπών είναι ένα πρώτο βήμα για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του από την αυτιλία. Γι' αυτό και έχουμε ολοκληρώσει την... Μάλλον θα ολοκληρώσουμε σχετική πρόταση πριν το καλοκαίρι. Ε, τώρα, διεθνεί διαπραγματεύσει ε, θα είμαι σύντομη, όχι γιατί δεν είναι σημαντικό, αλλά μπορούμε ίσω να επανέλθουμε κατά τη συζήτηση. Να σα πω ότι σε αυτή τη φάση πριν από το 2015 έχουμε πολλές ε, τύπες ε, ε, τυπικές επίσημες συνεδριάσεις, έχουμε και άτυπες όμως. Έχουμε το φόρουμ των μεγάλων οικονομιών, διπουργικές διμερείς, συζητήσεις ανάμεσα σε ένα σωρό περιφέρειες, και από αυτή την άποψη προχωράμε και στις επίσημες διαπραγματεύσεις στη Βόνη υπήρξε θετική ατμόσφαιρα, καθώς επίσης πιστεύω πως ε, ένα από τα πράγματα που βλέπουμε είναι πως αρχίζει να υπάρχει μια οικοδομητική συμβολή για το πώς μπορούμε πραγματικά να προχωρήσουμε όσον αφορά την μείωση του χάσματος όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει τη συμβουλευτική μας ανακοίνωση για τη Συμφωνία 2015 και θα καλωσορίζαμε οποιαδήποτε συμβολή. Γι' αυτό πολλοί από τους διεθνείς μας, διεθνείς μας εταίρους μιλούν για μια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω και είναι έτοιμοι να δουν τι κάνει ο καθένας. Από τη δική μου προοπτική εξακολουθώ να πιστεύω πως ένα από τα κύρια θέματα μέχρι το 2015 θα είναι ναι βέβαια χρειαζόμαστε πολύ προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και δραστηριότητα τέτοια, δεσμεύσεις. Αλλά μετά όταν θα έχουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και βλέπουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει κενό, πώς θα το καλύψουμε. Ποιο μπορεί να είναι το διαδικαστικό βήμα διεθνώς που θα προσθέσει κάτι ε, στην ύπαρξη διεθνούς πλαισίου. Είναι πολύ δύσκολη συζήτηση, αλλά και για τους πολίτες είναι μια από τις πιο σημαντικές συζητήσεις, γιατί αφορά το χάσμα φιλοδοξίας και το επίπεδο φιλοδοξίας. Για την ΚΟΠ νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι η φιλοδοξία πριν το 2020, πώς δηλαδή μπορούμε να προβούμε σε συγκεκριμένες συνεργασίες, σε διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίες, ανέφερα ότι τα φθοριούχα αέρια θα μπορούσε να είναι η μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, θα μπορούσε να είναι πάρκια σε ενέργεια, ορισμένοι μιλούν για συνεργασία για τα κτίρια. Ένα σωρό ιδέες κυκλοφορούν, αλλά αυτό που μπορούμε να περιμένουμε από τη Βαρσοβία είναι ίσως πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και τέλος, δύο ακόμα σημεία που είναι πολύ σημαντικά όσον αφορά την κόπτη της Βαρσοβίας, το ένα είναι η χρηματοδότηση. Και από την πλευρά της Κομισιόν είπαμε πολύ σαφώς στην Προεδρία της Λιθουανίας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να η Ευρώπη όταν θα φτάσει στη Βαρσοβία ε, και τα κράτη-μέλη θα έχουν κάποιες ιδέες για το πώς θα χρηματοδοτήσουν ε, το 14, το 15, το 16 κτλ. Στην πορεία προς το 2020 γιατί όλα αυτά σημαίνουν πολλά για τους φίλους μας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, αλλά και πολλά για την ψυχολογία ολόκληρη της διάσκεψης. Τέλος, να αναφέρω την επικύρωση, την επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιώτο. δουλεύουμε σκληρά γι' αυτό και να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, με μια παρατήρηση. Πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θα φτάσει η Ευρώπη στην Βαρσοβία ο υπόλοιπος κόσμος να μπορεί να δει πως ε, προχωράμε πολύ καλά στη διαδικασία επικύρωσης. Οι δικέ μου οδηγίε στι υπηρεσίε μου είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόταση από την Κομισιόν. Πιστεύω πω ε, όσο, όσο περισσότερο έχουν προχωρήσει τα κάτι σε αυτή την υπόθεση, τόσο καλύτερα. Και να πω και κάτι ακόμα, να σημειώσω ένα θέμα να το υπογραμμίσω. Νομίζω πω είναι λάθο αν στην Ευρώπη χρησιμοποιεί κανεί τη διαδικασία επικύρωσης, ώστε να γίνονται ένα σωρό εσωτερικέ συζητήσει για άλλα θέματα, ε, για παράδειγμα το μοίρασμα του βάρους ή για να προσθεθούν ε, πράγματα στους στόχους ε, του 2020. Αυτές οι συζητήσεις είναι ενδιαφέρουσες, αλλά δεν, έχουν, δεν είναι ο κατάλληλος χώρος η επικύρωση, γιατί ο υπόλοιπο κόσμος βλέπει, παρακολουθεί και αναρωτιέται, η Ευρώπη θα επικυρώσει αυτά, τα οποία, αυτά για τα οποία δεσμεύθηκε στην Τόχα ναι, το κάνουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να φανεί κιόλα πως κάνουμε τα απαραίτητα βήματα πριν φτάσουμε στη Βαρσοβία. Ja, vielen Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή Κόνη, βλέπουμε από την παρουσία σας ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να κάνουμε από το 2014 και επέκεινα. Το... Η κλιματική προβληματική λοιπόν δεν πρέπει να αφαιρεθεί από την πολιτική προβληματική. Έχουμε τον διάλογο τώρα με τους συντονιστές και πρώτος ο κύριος Ζέμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω και την Κόνη Χέντεγκάρ για την παρουσίασή της. Είσαστε ένας εξέχων εταίρος σε επίπεδο συνομιλιών πάντα κύριε Επίτροπε και γνωρίζουμε ότι για μας ως πολιτική ομάδα είναι σαφές ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε μια μόνιμη και βιώσιμη λύση στα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, να έχουμε μια αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τρόπο ο οποίος θα είναι και βιώσιμος και μόνιμος. Έχουμε κάποιες ανησυχίες για το θέμα της οπισθοφόρτησης του backloading, αλλά όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες επενδύσεις στις οποίες χρειάζεται η Ευρώπη στον τομέα αυτό. Αυτοί οι οποίοι θα επενδύσουν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μόνο με τον τρόπο θα μπορέσει να προχωρήσει η Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί λοιπόν για τα θέματα αυτά. Επίσης το ζήτημα με τα βιοκαύσιμα και τον παράγοντα ILUC, δηλαδή την αλλαγή, την επίπτωση της αλλαγής χρήσης γης, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία είδαμε ότι υπήρξαν ε, αρνητικά αποτελέσματα με την πρώτη γενιά βιοκαυσίμων και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Επίσης, ως ομάδα μας, έχουμε, ως ομάδα του ΕΛΚΑ, έχουμε καταθέσει μια σειρά τροπολογιών. Τώρα πώς θα γίνει η ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια αυτό θα το δούμε στην πράξη. Αλλά ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και θέλω να επιχειρηματολογήσω και πάλι ενώπιον σας κυρία Επίτροπε ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα μοντέλα για να αντιμετωπίσουμε τις εκπομπές από την αυτιλία και από τον αεροπορικό κλάδο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μέχρι το 2020 ώστε όσο δυνατόν ε, περισσότερο να φέρουμε αυτούς τους τομείς μέσα σε ένα νέο σύστημα και το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει θέσει φιλόδοξους στόχους δεν θα πρέπει να οδηγήσει και σε μετακίνηση όλων των βιομηχανικών κλάδων από την Ευρώπη. Θα πρέπει να σκεφτούμε για το θέμα των στόχων στο κλίμα, αλλά και σε ό,τι αφορά το τίμημα της ενέργειας. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά με ένα βιώσιμο τρόπο. Εμείς σας στείλουμε χείρα βοηθεία από την πλευρά του ΕΛ και σα ζητούμε να έχετε πάντα υπόψη σας την ανάγκη να υπάρξει και προστασία του περιβάλλοντο και τη αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή, αλλά να έχουμε και ένα κλίμα το οποίο θα παραμείνει ευνοϊκό και θετικό για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και όχι εχθρικό. Και ελπίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε τη συνεργασία στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, <laughs> έχετε υποστηρίξει πάρα πολλά. Αυτό το οποίο δεν ξέρει κανεί είναι πώς θα πάει η ψηφοφορία για τους σοσιαλιστές, η Λίντα Μακάβεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Έχετε την υποστήριξη της σοσιαλιστικής ομάδας για να μπορέσει να υπάρξει κάποια λύση για την οπισθοφόρτηση. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα πείσουμε τους συναδέλφους που δεν υποστήριξαν αυτό το μέτρο την προηγούμενη φορά. Αν θέλουμε να πάμε σε διεθνείς συνομιλίες, όπως είπατε, θα είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό αν καταρρεύσει το ETS, το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Μιλάμε για το τι θα κάνουμε με τις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου στο μέλλον, αλλά αν δεν περάσει αυτό το, μέλλον, το μέτρο και δεν έχουμε άλλες λύσεις εκτός από το ETS. Τα προβλήματα του ETS δεν μπορεί να είναι η δικαιολογία να μην αντιμετωπίσουμε τώρα τα προβλήματα που έχουμε αν δεν τα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, δεν θα υπάρχει το σύστημα εμπορία εκπομπών, ώστε να μπορούμε να το μεταρρυθμίσουμε στη συνέχεια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αντίπαλα συστήματα, όπως αυτό το Αυστραλιανό. Θα πρέπει να δώσουμε στους αντιπάλους μας τη δυνατότητα να νομίζουν ότι κερδίζουν, το επιχει... κερδίζουν την το διάλογο αυτή τη στιγμή, ότι προχωρούν. Θα πρέπει να είμαστε σαφεί σε αυτά τα οποία προσπαθούμε να επιτύχουμε σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι προσπαθούμε να επιτύχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λέτε, κύριε Επίτροπε, ότι αυτή τη στιγμή μερικέ φορέ είναι πάρα πολύ δύσκολο σε όλα αυτά τα μεγάλα θέματα για το θέμα του ILUC. Ακούμε τι προτάσει από το Συμβούλιο κτλ. Πολλέ φορέ είναι αρνητικά, αλλά διάβασα στου Financial Times χθε ότι οι Κινέζοι εξετάζουν πάρα πολύ προσεκτικά και σοβαρά το να περιλάβουν και στόχους μείωσης των εκπομπών στο επόμενο πενταετές του σχέδιο ανάπτυξης. Και βλέπουν για τον ορίζοντα του 2016-2020 μέτρα για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Αν οι Κινέζοι πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, και στις ΗΠΑ βλέπουμε να υπάρχει περισσότερη ενεργητικότητα για τα θέματα αυτά και πιο πολύ κίνηση προς τις ανανεώσιμες ενέργειες. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία και για μας να πάμε στις διεθνείς συνομιλίες με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Θα ήθελα να μου πείτε κάτι για τους ασφαλτικούς, ασ, τις ασφαλτικές άμμους και την εξόρυξη πετρελαίου από αυτές. Και υπάρχουν επίσης και συζητήσεις οι οποίες ξεκινούν για τη χρήση της βιομάζας. Υπήρξαν προβλήματα με το με την επίπτωση στο κλίμα από την αλλαγή χρήσης γης στο Άιλουκ και τώρα που τα βιοκαύσιμα έχουν περάσει σε δεύτερη φάση έχουμε τη συζήτηση για τη βιομάζα. Ξέρω ότι τα θέματα αυτά τα αντιμετωπίζει η Κομισιόν σαν σύνολο και όχι μονάχα η υπηρεσία σας αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε αν θέλουμε να και με ξύλα στους σταθμούς ενέργειας και αν το κάνουμε αυτό ποια είναι τα κριτήρια βιωσιμότητας και πολλοί βιομηχανικοί κλάδοι θέλουν να εξασφαλίσουν ότι υπάρχουν εδώ τα κριτήρια βιωσιμότητα, δεν θέλουν να κάνουν επένδυση σε χρήση βιομάζα για ενέργεια και μετά να δούνε ότι όλα αυτά θα σταματήσουν απότομα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σαφήνεια και χρειαζόμαστε αυτή τη σαφήνεια το ταχύτερο δυνατό. Αλλιώ μπορούμε να επαναλάβουμε τα ίδια σφάλματα που έγιναν με τα βιοκαύσιμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Κρι επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε θα σας ρωτήσω κάτι δύσκολο, αδύνατο σχεδόν. Ε, το μεσημέρι μίλησα σε μια συνεδρίαση για τεχνολογίες εκπομπών, χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Και πραγματικά, εάν θέλουμε να δώσουμε στην βιομηχανία πραγματικά κίνητρα για επενδύσεις του άνθρακα. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια καλή τιμή άνθρακα, γι' αυτό και χρειαζόμαστε το backloading και σε αυτό το κοινοβούλιο βέβαια και στο Συμβούλιο υπάρχει ανησυχία για το ότι θα χαθούν δουλειές ενδεχομένω και αυτό πιέζει τη βιομηχανία. Και αυτό δημιουργεί εμπορικό μειονέκτημα στην Ευρώπη και μια γενικότερη καχυποψία ότι δεν θα καταφέρουμε από το 2015 και μετά να επιτύχουμε τους στόχους μας. Πώς μπορεί λοιπόν το Συμβούλιο να κερδίσει. Το backloading είναι μόνο ένα πρόβλημα, η τεχνητή απόσυρση δικαιωμάτων δηλαδή. Την περασμένη εβδομάδα άκουσα ότι ο Γενικός Διευθυντής της ε, Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος διοχέτευσε πιστοποιητικά στην αγορά έτσι ώστε να τονώσει τις επενδύσεις στην ε, στις τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Θα ήθελα να μάθω από πού προέρχεται αυτή η εντολή. Ευχαριστώ πολύ, Ήβης, για τις ερωτήσεις. Σαν του χάσει, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την Επίτροπο που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Ένα πιο γενικό ερώτημα για αρχή. Αναφέρεται τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην πρόσφατη διάσκεψη σε την ε, πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ε, στόχους για το 2030. Δεν θα έπρεπε όμως να χρειαζόμαστε ήδη νομοθετικές προτάσεις μέχρι το τέλος αυτού εδώ του χρόνου για το 2030, διότι εάν δεν έχουμε κάποια νομοθετική πρόταση, η αυτή η ασάφεια θα επιμείνει μακροπρόθεσμα. Και η αγορά του άνθρακα μας δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται φύση κανόνες για να παίξουν. Επίσης, αυτά όσον αφορά τα διαρθρωτικά προβλήματα στο σύστημα εμπορία εκπομπών. Και τώρα κάτι πιο συγκεκριμένο. Αναφέρεται τους στόχους διοξιδίου του άνθρακα για τα οχήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να υπάρχουν όρια για το 2025. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει την πρόταση αυτή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πιστεύω πως αυτός θα ήταν ένας αποδοτικότερος τρόπος για να δείξουμε στην αυτοκινητοβιομηχανία την κατεύθυνσή μας εν ώψη της επόμενης πρότασης τα επόμενα χρόνια. Και επίσης, τι γίνεται με τις εκπομπές των πλοίων. Η τελευταία απόφαση είχε ως εξή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπέβαλε πρόταση στο πρώτο μισό αυτού του χρόνου. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω πού βρισκόμαστε. Και κάτι τελευταίο, όχι τόσο ερώτηση, μια παρατήρηση σχετικά με τον ε, Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. έχει παρατηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ευρωπαϊκή προσέγγιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών σε μεγάλες αποστάσεις, σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Έχει υποχωρήσει δηλαδή απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείες, οι οποίες έχουν μία προσέγγιση περισσότερο εναερίου χώρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, σαν του χάσει. Με εσάς ολοκληρώθηκε ο γύρος των συντονιστών. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Επίτροπο έτσι ώστε να απαντήσει τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ξεκινώ με τα τελευταία ερωτήματα. Η Κομισιόν δεν θα σταματήσει τις προσπάθειές της σε οποιοδήποτε θέμα. Η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί να κάνει μαζί με τα κράτη-μέλη για να βρει ένα καλό τρόπο να προχωρήσουμε για τα θέματα αυτά. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Δεν ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να βρούμε συμμάχους για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι πετυχαίνουμε κάποια πρόοδο, εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα από όλη αυτή τη διαδικασία του ικανοτορασμού πολιτικής αεροπορίας σε διεθνές επίπεδο, αλλά πρέπει να πω ότι και οι ομόλογοι μας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δείξουν σοβαρότητα. Δεν τους άρεσε το ευρωπαϊκό περιφερειακό σύστημα. Ίσως θέλουν ένα παγκόσμιο σύστημα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόματα. Θα πρέπει αυτοί να αρχίσουν να αλλάζουν τις θέσεις τους για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο σύστημα και να κάνουμε όλοι κάποιους συμβιβασμούς προς την κατεύθυνση αυτή για τον Ρίτσαρτ Ρίχαρτ Ζέμπερ και τη Λίνα Μαγκάβεν για το θέμα της οπισθοφόρτησης. Το το οποίο βλέπω είναι μια θέληση να αναζητηθεί μια συμβιβαστική λύση και θα ήθελα να ξέρω ότι θα προκύψει βέβαια από την εσωτερική διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις ψηφοφορίες. Νομίζω ότι όλα αυτά θα είναι πολύ θετικά, όπως προσπάθησα να είμαι σαφής. Είμαστε απόλυτα ανοιχτοί να συμπεριλάβουμε και νέες ιδέες εάν διατυπωθούν η Λίνα Μακάβεν ρώτησε για την Κίνα. Νομίζω ότι ήδη μέσα σε αυτό το τρέχον πενταετέ σχέδιο η Κίνα έθεσε κάποιους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το καινούριο στοιχείο είναι όμως είναι ότι η βάση των ε, δηλώσεων κάποιων υψηλών αξιωματούχων και αυτό περιλαμβάνει και κάποιους ερευνητές το νέο στοιχείο της Εθνικής Επιτροπής ε, Ανάπτυξης είναι το ερώτημα του αν θα πρέπει να θέσουν ένα ανώτατο όριο στις ε, εκπομπές και αν θα πρέπει να υπάρξει εμπροστοφόρτιση για τα έτη εχμής, να υπάρξει δηλαδή κάποιο όριο με τα χρόνια όπου θα κορυφωθούν οι εκπομπές. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα προκύψει και εγώ βλέπω και τις εκθέσεις που προέρχονται από το εσωτερικό της Κίνας. Δεν ξέρουν πολύ περισσότερο από ό,τι ξέρουμε εμείς από τα μέσα ενημέρωση. Πιστεύω όμως ότι αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι εκεί βρίσκονται τα πραγματικά ερωτήματα. Αυτά είναι τα δύο κέρια ερωτήματα για την Κίνα. Πότε θα πρέπει να φτάσουν σε, στο ανώτατο σημείο οι εκπομπές τους και αν θα εφαρμόσουν μια οροφή. Έχουν ξεκινήσει την, την εμπορία εκπομπών, το ξεκινήσανε στην Σανκάη και στο Τσιν Θα μπορέσουν λοιπόν να τεθούν σε εφαρμογή και περισσότερα σχέδια αυτού του είδους και θέλουν ήδη για το 2016 να έχουν ένα εθνικό σύστημα που να καλύπτει όλη την Κίνα για εμπορία εκπομπών. Αυτό λοιπόν μπορεί να αποβεί πολύ ενδιαφέρον. Για τις ε, ασφαλτικές άμμους η έκθεση αντικτύπου δεν έχει ακόμα περατωθεί, θα την έχουμε το καλοκαίρι ή αργότερα. Chris Davis, ακόμα και οι γενικοί διευθυντές μπορεί καμιά φορά να σκέφτονται αυθόρμητα. Αυτή ήταν μια ιδέα που ήρθε κάπως απρόοπτα. Ήταν κάτι το οποίο όμως είχε ήδη ε, αντιμετωπιστεί στην διαδικασία διαβούλευση γιατί πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι είχαν καταλήξει σε παρόμοιες ιδέες. Σας υπενθυμίζω κάναμε τη δεύτερη ε, πρόσκληση για το NER 300 πιο νωρίς από ό,τι προβλεπόταν και γίνεται τώρα την πρώτη, την πρώτη του Ιουλίου θα είναι η καταληκτική προθεσμία για αυτή τη δεύτερη πρόσκληση. Ποια είναι η κατάσταση στο Συμβούλιο για την Οπισθοφόρτιση. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρετε ήδη. Ήταν ενδιαφέρον αυτό το οποίο ακούσαμε από τη γερμανική ηγεσία σε μια δημόσια συνδιάσκεψη ότι και η Καγκελάριος θα υποστήριζε τις διαθροντικές επιλογές, την οπισθοφόρτιση για την αγορά άνθρακος. Ήταν επίσης όμως σαφές ότι θα ήταν πιο εύκολο να γίνει αυτό μετά από τις γερμανικές εκλογές από ότι πριν από τις γερμανικές εκλογές. Από αυτά που γνωρίζω με τις επαφές που έχουμε με τις διάφορες κυβερνήσεις, υπάρχει μια σημαντική πλειοψηφία κυβερνήσεων που υποστηρίζει την οπισθοφόρτηση, αλλά ξέρουμε όλοι που, βρίσκεται, που βρίσκονται τα προβλήματα και νομίζω ότι αναπόκειται και στην Ιρλανδική Προεδρία να απαντήσει ερωτήματα για το πότε το Συμβούλιο θέλει να προχωρήσει σε πιο επίσημο επίπεδο για να γίνει μια ψηφοφορία στο Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Στην ΣΑ του Χάση οι νομοθετικές προτάσεις για το 2030. Όταν συζητήσουμε το 2030 και την πράσινη βίβλο στην Κομισιόν, όταν το συζητήσαμε μάλλον, δεν είχε αποφασιστεί ακριβώς Είχαμε πει ότι το επόμενο βήμα θα πρέπει να γίνει πριν από το τέλος του χρόνου, αλλά αν θα είχε το χαρακτήρα νομοθετικής πρόταση ή κάτι άλλο, αυτό δεν είχε αποφασιστεί. Επομένω δεν είχε υπάρξει μια απόφαση από την Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι αργή κάτω και κυβερνήσεων είπαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θέλουν απλώ μια πρόταση ή μια νέα βίβλο, πράσινη, άσπρη, οτιδήποτε. Θέλουν συγκεκριμένε προτάσει. Γι' αυτό ξέρω ότι οι συνάδελφοί μου στην Κομισιόν θα προσπαθήσουν να δώσουν κάποια απάντηση και κάποια συνέχεια σε όλα αυτά. Αναφερθήκατε <laughs> για το στόχο του 2025 για τα οχήματα, για τα αυτοκίνητα. Η Κομισιόν πιστεύει ότι πράγματι πρέπει να δώσει στην βιομηχανία ένα ορίζοντα για τη σχεδίαση, όπως λέτε, και πάντα μια πρώιμη αναθεώρηση είναι καλύτερη από μια ε, εκ των υστέρων αναθεώρηση όταν ξέρει κανείς, μια όψιμη αναθεώρηση όταν ξέρουμε πώς ε, πόσο μεγάλο είναι ο κύκλο ε, ανάπτυξη τη βιομηχανία. Υπάρχουν ορισμένε κυβερνήσει οι οποίε θα προτιμούσαν μια όψιμη ε, αναθεώρηση. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει κανεί με όλα αυτά, αλλά μα ενδιαφέρει να μπορέσουν οι βιομηχανίε να προσαρμοστούν σε ένα κύκλο ε, παραγωγή ο οποίο είναι τη τάξη των 7 ετών. Και αυτά τα οποία είναι τώρα στα εργαστήρια είναι τα αυτοκίνητα τα οποία πολύ σύντομα θα βρίσκονται στον οριζόντα μετά το 2025. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε με τα θέματα αυτά, τόσο καλύτερα. Αυτά. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο γύρο. Πέτερ Λίζε, Τζο Λάινεν. Υπάρχει κάποιος άλλος τον οποίον τον λησεμόνισε. Όχι. Μπορώ να κλείσω λοιπόν τον κατάλογο. Ο Μιλτών δίνω το λόγο στον Πέτερ Λίζε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Πίτροπο. Θα ήθελα να σταθώ στο τελευταίο θέμα με το οποίο εσείς κλείσατε την ομιλία σας. Τα οχήματα και τους, ε, τις προδιαγραφές για την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος στον οριζόντα το 2025. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια ευρεία πλειοψηφία στην ε, Επιτροπή μας, ώστε να έχουμε την πλειοψηφία αυτή για τους στόχους του 2025. Αυτή τη στιγμή ο συγητής μας διαπραγματεύεται με το Συμβούλιο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν υπάρξει μια πρόταση της Κομισιόν να συμπεριληφθεί στη διαδικασία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ έχω δει τα τελευταία χρόνια ότι μπορούσαμε να έχουμε ε, κάποιες ε, συμφωνίες εγκαίρως και κατά τη δική μου άποψη οι, οι στόχοι που έχει ενδεικτικά εγκρίνει η Επιτροπή μας για τις εκπομπές δεν είναι τόσο μακριά από αυτά που έχουν αποφασιστεί μόλις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει και μια πολύ επίκαιρη συζήτηση για τον κύκλο δοκιμασίας για τα οχήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον καταναλωτή και φυσικά ενδιαφέρει και το περιβάλλον, την προστασία του περιβάλλοντος. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη διάσταση μεταξύ της πραγματικής κατανάλωσης και των πραγματικών εκπομπών και αυτών οι οποίες παρουσιάζονται ως πρότυπα από τους βιομηχάνους. Αυτό σημαίνει ότι ο κύκλος αυτός δοκιμασίας δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα και θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αν μπορεί και ο ειδικό μα εισηγητής μα να υποστηρίξει την κίνηση προς μια διεθνή μεταρρύθμιση των ε, κύκλων δοκιμασιών για τα οχήματα, γιατί αυτό ενδιαφέρει και το περιβάλλον, αλλά και ενδιαφέρει και τους ε, καταναλωτές οι οποίοι θέλουν να βασίζονται στις ε, τιμές που τους δίνουν οι βιομηχανίες. Για το σταμάτημα του ρολογιού, εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν να μην βρεθούμε σε μια θέση η οποία θα είναι αρνητική για μας. Η εντύπωση <clears throat> του κοινού είναι ότι φεύγει η βιομηχανία και πηγαίνει στην Κίνα, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν δεν τους κάνουν τα χατηρία, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε τις διαπραγματεύσεις και να εξασφαλίσουμε ότι θα, <clears throat> θα υπάρξει κάτι που θα ακολουθήσει το πάγωμα του ορολογιού για ένα χρόνο από την ΙΚΑΟ. Κύριε Επίτροπε, σύμφωνο ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για το περιβάλλον τώρα σε περίοδο οικονομικής κρίσης και έχουμε πάρει λάθος δρόμο πιστεύω όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ στην Ευρώπη έχουμε την ευκαιρία πραγματικά να χαράξουμε οικολογική βιομηχανική πολιτική και μάλιστα καλή, αλλά αυτό που με ανησυχεί, ιδιαίτερα με την τελευταία διάσκεψη κορυφής για το κλίμα, είναι ότι έγινε μια μαζική επίθεση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Επιτροπή. Το επιχείρημα ήταν ότι είναι πολύ ακριβές αυτές οι πηγές ενέργειας. Και πραγματικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε να προστατεύσουμε αυτές τις ανανεώσιμες πηγές. Έχουν επενδυθεί πάρα πολλά κονδύλια και διακυβεύονται πάρα πολλά. Όσον αφορά το σύστημα εμπορία εκπομπών, πράγματι προσπαθούμε σε δεύτερο κύκλο να προχωρήσουμε με το backloading, με την οπισθοφόρτιση. Όντως υπάρχουν προβλήματα. Αυτό που έχω παρατηρήσει όμως είναι ότι η βιομηχανία δεν έχει προβλήματα με αυτό και μας ρωτά τι γίνεται στη συνέχεια, τι θα γίνει μετά το 2020, ποιες θα είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές που θα γίνουν. Και πραγματικά υπάρχει εδώ ένα νευραλγικό σημείο όσον αφορά την, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και παρατηρώ ότι η προσφορά όλο ένα και μεγαλώνει. Και αυτό επηρεάζει το σύστημα. Ίσως θα μπορούσατε εσείς να μας πείτε λεπτομέρειες. Τώρα, όπως είπε και η ΣΑ του Χάση για τους στόχους του 2030, βρισκόμαστε όντως σε προεκλογική περίοδο και πρέπει πραγματικά να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θα βοηθήσει καθόλου την προεκλογική μας περίοδο και οι μεγάλοι επενδυτές μας το θεωρούν πολύ σύντομο αυτό. Την ε, περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο, με μεγάλο κόπο, ψηφίσαμε την ε, συνέχιση του ε, στόχου της ενεργειακής απόδοσης, τη δρομολόγησή του. Τώρα, όσον αφορά τα οχήματα, ήμουν στην διάσκεψη για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα στο Βερολίνο ο στόχος είναι το 1 εκατομμύριο ηλεκτρονικά αυτοκίνητα μέχρι το 2020. Είμαι πιο φιλόδοξος, ελπίζω σε περισσότερα, σε 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα, αλλά εδώ για να το επιτύχουμε αυτό χρειαζόμαστε μια νέα μέθοδο ελέγχου των εκπομπών και της μέτρησης των εκπομπών των οχημάτων αυτών. διότι στην επιλογή του παρόχου ενέργειας οι εκπομπές είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάινεν, Μπάς Άικχαουτ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και την Επίτροπο Χέντεκαρτ για την εισαγωγή της. Δεν θα επιχειρηματολογήσω για το backloading. Έχουν ήδη ακουστεί τα επιχειρήματα. Προχωράμε προς συμβιβασμό και να ευχαριστήσω εδώ τον Ρίχαρτ Τζέιμπερ για την προθυμία του για συμβιβασμό. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αυτό που θα ήθελα, κυρία Επίτροπε, να σας ε, ρωτήσω είναι για κάποια άλλα ζητήματα. Καταρχάς, να απαντήσατε στην ερώτηση της Ελίντα για τη βιομάζα, για τα μη βιώσιμα κριτήρια για τη βιομάζα. Εάν δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη το χρέος, το έλλειμμα που έχει η βιομάζα σε άνθρακα, πρέπει να δούμε ότι αυτό είναι κάτι προβληματικό. Είναι κάτι που χρειαζόμαστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κολλησιαρχεί. Τώρα, ένας άλλος επίτροπος, ο οποίος ε, είναι ο Επίτροπος Ταγιάννη και ασχολείται με πολύ ενδιαφέροντες φακέλους, τον Ιούνιο θα προτείνει ένα ατσαλένιο σχεδίο δράσης. Και στα πλαίσια αυτού του σχεδίου δράσης θα ακούσουμε προτάσεις για την βιομηχανία λοιπόν χάλιβα. Έχουν λάβει αυτές οι βιομηχανίες λοιπόν δωρεάν πιστοποιητικά. Και δεν θέλω πραγματικά να ακούσω ε, επιχειρήματα του τύπου το ETS, το σύστημα εμπορία εκπομπών, σκοτώνει τη βιομηχανία χάλιβα. Αυτά είναι ανοησίε. Όπως επίσης ότι δεν υπάρχει καμία άνθηση της ε, οικονομίας ε, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Και να πω ότι πραγματικά η μόνη ευκαιρία για άνθηση οικονομίας είναι στον κλάδο των ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας. Και χρειάζεται λοιπόν μια σωστή τιμολόγηση των εκπομπών άνθρακα για να καρποφορήσει αυτή η βιομηχανία. Τελευταίο ζήτημα. Ένας επίτροπος από τον οποίο περιμένω δράση. Αναφέρομαι στην Γενική Διευθυνσία Ανταγωνιστικότητας. Αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται ένα σύστημα τιμών για 40 χρόνια για την πυρηνική ενέργεια, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή τη στιγμή συζητά μία εγγύηση τιμών για την πυρηνική βιομηχανία για τα επόμενα 40 χρόνια. Και αυτό πραγματικά είναι ό,τι πιο ανόητο μπορεί να κάνει κανείς. Και σας διαβεβαιώ ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνιστικότητας θα επιληφθεί άμεσα του θέματος και πραγματικά ελπίζω εσείς να ασκήσετε πίεση στους συναδέλφους σας έτσι ώστε αυτή η ανοησία να μην λάβει χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος συνάδελφος ο κύριος Μπόρισλαβ Σόνικ. Ε, κυρία Επίτροπε, για το backloading, την καθυστέρηση Νομίζω πως βλέπουμε δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Ε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά τον Απρίλιο το Κοινοβούλιο είπε όχι σε αυτή την καθυστέρηση και τώρα ξανάρχεται με σχεδόν ένα στρατιωτικό τρόπο, λες και είναι να υπογράψουμε κάποια συμφωνία ειρήνης. Δεν νομίζετε πως είναι κάπως προσβλητικό για το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις και το δέχεστε, αλλά τελικά συνεχίζετε να επανέρχεστε μέχρι ότου πετύχετε αυτό που θέλετε. Μάλιστα αυτή η πρόταση πραγματικά καταψηφίστηκε στην Επιτροπή. Ισχύει. Στο τέλος της πρώτης ανάγνωσης δεν είχαμε καμία πλειοψηφία. Έτσι προς ενημερωσή σας, η Ολάντα Χιπνέρ, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο προηγούμενος ομιλητής. Επίτροπε, γιατί δεν αποσύρετε την πρότασή σας. Η παροχή μειώθηκε, η προσφορά μάλλον ε, μειώθηκε και δεν ε, μπορεί να σωθεί η κατάσταση μέσω της καθυστέρησης ή του backloading. Γνωρίζουμε πως εάν αυτό δεν επιτύχει θα προσφερθούν νέες διευθυντικές πληροφορίες. Εμείς δεν έχουμε λάβει καμία σχετική ενημέρωση και το Κοινοβούλιο συμφώνησε να μην κάνει καμία τεχνητή παρέμβαση στην αγορά. Ωστόσο κάποιοι λένε τώρα πως το backloading ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να προστατευτεί το περιβάλλον. Τον Απρίλιο, όταν ε, συναντηθήκαμε, είπατε ότι η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρώπη θα, κατά 20% θα είχε επιτευχθεί μέχρι το 2015. Έγινε κάτι το μεταξύ τους δύο τελευταίους μήνες. Μπορείτε να μας πείτε κάτι ε, κάποια έρευνα, κάποια πορίσματα ερευνητικά που θα μας πείσουν ότι δεν θα καταφέρουμε αυτό το στόχο. Γιατί με κάποιο τρόπο θα πρέπει και εμείς να διαβάσουμε αυτές τις πληροφορίες στους ψηφοφόρους μας. Η απόφαση του Κοινοβουλίου ήταν αρκετά ξεκάθαρη. Εμείς καταλέξαμε στο, ότι το backloading ήταν υπερβολικά, υπερβολική παρέμβαση στην αγορά. Τι θα μας πείτε αν τελικά αποδειχθεί ότι το Κοινοβούλιο για δεύτερη φορά θα απορρίψει την πρόταση αυτή. Θα την ξαναυποβάλλετε τρίτη φορά ή πιο συγκεκριμένες και διαφορετικές προτάσεις για το 2020. Ευχαριστώ πολύ. Κρίστα Κλάς, επόμενη ομιλήτρια. Αυτό που είπε η Γιολέντα Χιούπνερ για το backloading ισχύει για την οδηγία για τη βιομάζα και πρέπει να δούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με, μάλιστα με πολύ μεγάλη προσοχή. Θα ήθελα να αναφερθώ στα βιοκαύσιμα. Μα είπατε ότι τα βιοκαύσιμα πρέπει να είναι βιώσιμα. Αυτό το συμμερίζομαι απόλυτα. Τα κριτήρια της βιωσιμότητας όμως, ιδιαίτερα όσον αφορά τα, ε, τις τρίτες χώρες, πρέπει να είναι σαφή. Υπάρχουν προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Αγεωργίας, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν τώρα. Μιλήσατε για μία μελέτη, η οποία δεν έχει τύχει μεγάλη στήριξη, διότι αναφέρονται πολιτικά κίνητρα και δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν καινοτομίες. Διάβασα για παράδειγμα πρόσφατα ότι στην Γερμανία οι καλύτερες ε, καινοτομίες όσον αφορά την βιομάζα βραβεύονται. Δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα επιβράβευσης λοιπόν καινοτόμων τεχνολογιών. Αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε, να το προωθήσουμε, να δούμε τους επιμέρους παράγοντες οι οποίοι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να έχουμε τις ε, νεότερες και πιο σύγχρονες ε, τεχνολογίες. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα κάθε χρόνο να υπολογίζουμε το επίπεδο εκπομπών μας και να κάνουμε προβλέψεις και για την ε, έμεση χρήση της γης. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ναι, Γιόργενσεν, έχετε το λόγο τελευταίος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Επίτροπε. Όταν συζητάμε το backloading, ένα από τα αρνητικά σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε το παράδειγμα στους υπολείπους, στον κόσμο. Πώς θα δώσουμε το παράδειγμα άμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ στην Ευρώπη εμείς. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν ποιες ήταν οι αντιδράσεις ε, των ε, ομολόγων σας στα άλλα μέρη του κόσμου και τι περιμένουν να γίνει στην Ευρώπη. Έπειτα Αναφέρατε τη στρατηγική που θα πρέπει να έχουμε ως ε, Ένωση πριν από την ε, συνεδρίαση στη Παρίσι και μετά στην Βαρσοβία. Ε, αυτό λέμε βέβαια κάθε χρόνο, τα όσα είπατε εσείς. Και κάθε χρόνο μόλις εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μιλάμε μια φωνή. Πολύ συχνά, πάση περιπτώσει. Ίσως λοιπόν αυτή τη φορά να υιοθετούσαμε μια άλλη στρατηγική, όπου όντως θα μιλήσουμε με μια φωνή. Και μια λύση για να το κάνουμε αυτό είναι πολύ απλή, να πιέσουμε το Συμβούλιο ώστε να αρχίσει να παίρνει αποφάσει ψηφίζοντας. Γιατί όλες οι χώρες πρέπει κάθε φορά να συμφωνούν για τα πάντα. Δεν το κάνουμε αυτό για άλλα πολιτικά θέματα. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου μια χώρα έχει μπλοκάρει ε, τη δυνατότητα εξέλιξης μιας ε, υπόθεσης για χρόνια. Αυτό πρέπει πια να σταματήσει. Και έπειτα, ποια είναι η θέση σας όταν σας ρωτούν αν θα πρέπει να μείνουμε κάτω από τους δύο βαθμούς. Μιλάμε για στρατηγικές, για νομοθεσία, μα εδώ μιλάμε και για να σώσουμε το κλίμα. Και από όσο γνωρίζω, οι πολιτικές μας ε, βασίζονται στους υπολογισμούς των Ηνωμένων Εθνών και λένε ότι οι δύο βαθμοί θα, θα βγουν όταν θα είμαστε στα 500 ppm, ενώ αν δεν αλλάξουμε τώρα θεμελιωδώς, αν δεν αλλάξουμε βασικά ρηξικέλευτα την τακτική μας, ε, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσουμε. Τι λέτε εσείς λοιπόν όταν σας ρωτάνε αν μπορούμε να σταθεροποιήσουμε τους δύο βαθμούς. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν και αυτό τον κύκλο. Έγινε πιο σύντομα από ό,τι περίμενα. Τόσο λίγες λέξεις λοιπόν από την παρουσίασή σας προκάλεσαν τόσες πολλές ερωτήσεις. Βλέπετε και εδώ και στην Ολομέλεια. Η πρόταση για το backloading δεν έχει απορριφθεί τελείως αλλά έχει παραπέμφθει για επανεξέταση. Θα δούμε τι θα γίνει στην δεύτερη πληροφορία, στην πρώτη δεν είχαμε πλειοψηφία. Είναι κάτι φυσιολογικό. Θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε δεύτερη ανάγνωση. Και αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε την πρόταση έτσι ώστε να πείσουμε εκείνους που την απέρι... απέριψαν τουλάχιστον να τους κάνουμε να το ξανασκεφτούν και να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε κάποιον συμβιβασμό. Είναι λοιπόν πραγματικά συναρπαστικές αυτές οι στιγμές θα έχουμε πολύ παραγωγικούς επόμενους μήνες. Όπως είπε και ο συνάδελφος, περιμένουμε ένα σχέδιο δράσης για τον Χάλιβα. Ή ο κλάδος ε, της αιωλικής ενέργειας είναι ο δεύτερος ο μεγαλύτερος αγοραστής λοιπόν προϊόντων Χάλιβα. απασχολεί πάνω α, απασχολεί δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους Χρειαζόμαστε λοιπόν την βιομηχανία την Ευρω... στην Ευρώπη. Βιομηχανία που καταφέρνει να προσελκύσει όλο και περισσότερους εργαζομένους ή να μεταφέρει εργαζομένους από τομέα σε τομέα. Δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα η άσπρα, η μαύρα, κακούς και καλούς. Η βιομηχανία πραγματικά διασφαλίζει την ευημερία μας. Και πρέπει να βρούμε τα κοινά σημεία παρά να τονίσουμε τις διαφορές. Θα δώσω τώρα το λόγο για τα τελικά σας σχόλια, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Έχει φύγει ο Πιτέρα. Λίζε, έχω κάνει κάποια σχόλια για τα α, οχήματα είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω να υπάρξει ένα σαφέ μήνυμα προ την αυτοκινητοβιομηχανία για τον Γιώ Υπάρχει η θέληση να υπάρξουν στόχοι για το 2030 πριν από τις ευρωεκλογέ του χρόνου. Με τον τρόπο που εγώ το ερμηνεύω αυτό, τα συμπεράσματα μάλλον που ερμηνεύω τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι είναι σαφέ ότι θέλουν να επανέλθουν στο θέμα αυτό το Μάρτιο του 2014. Γι' αυτό υπάρχει μια σαφή σύνδεση, ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Δεν πρέπει να αυταπατώμεθα αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν για τα θέματα αυτά και για λόγους του ενεργειακού τομέα και της βιομηχανίας θα πρέπει να έχουν μια καλύτερη γνώση προς τα που πηγαίνουμε. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να είναι μια εύκολη συζήτηση στο Συμβούλιο δεν είναι ότι επειδή δώσαμε σημασία στο θέμα αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε το αν θα επιταχύνουμε ή όχι τον καθορισμό των στόχων για το 2030. Είναι σαφές ότι μέσα στους επόμενους δέκα μήνες τα κράτη, οι αρχηγοί των κρατών μελών θέλουν να επανέλθουν στο θέμα αυτό και αυτό θα προσδιορίσει και το έργο της Κομισιόν. Σε εσωτερικό επίπεδο μιλήσατε για τις διαφορετικές επιλογές σε σχέση με το 2030. Είναι σαφές όταν είχαμε αυτή την πρώτη διτή προσέγγιση Θέλαμε να έχουμε πιστοφόρτιση για να σταθεροποιήσουμε το σύστημα, ενώ προσπαθούμε να εξετάσουμε τι πιο φιλόδοξε διαρθωτικέ επιλογέ. Τώρα βλέπετε για λόγου που ξέρουμε όλοι ότι έχει υπάρξει μια αναβολή όλων αυτών. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Η πραγματικότητα είναι ότι η συζήτηση για τις πιο διαρθρωτικές επιλογές θα συμπέσει και θα συμβάλλει με τη συζήτηση για το 2030. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν τελικά ποιο θα είναι το σύστημα τιμολόγησης και ποιοι θα είναι οι στόχοι για το 2030 στην Ευρώπη. Υπάρχει κάτι το οποίο για μένα είναι αξιοσημείωτο. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε τις ε, συστάσεις αναχώρα σήμερα για, μια, για κάθε μια από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και μια ανακοίνωση όπου λέει ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό είναι η κυριότερη προτεραιότητά μας στην Ευρώπη. Και λέει αυτή η ανακοίνωση ότι η δυνατότητα δημιουργία θέσεων απασχόληση τη πράσινη οικονομία δεν έχει ακόμα τύχη πλήρου εκμετάλλευση. Και υπάρχει μια ισχυρή διατύπωση που να τονίζει γιατί τα κάτι μελη θα πρέπει να κάνουν κάτι περισσότερο για την αξιοποίηση των πόρων με αποτελεσματικό τρόπο, την αποδοτικότητα της ενέργειας, τη χρησιμοποίηση μιας οικονομίας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και πάλι προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τα κάτι μελη να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση, καμία αντίφαση μεταξύ του να κάνουν μια ευφυά πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και συγχρόνως να αντιμετωπίζουν την έλλειψη θέσεων απασχόλησης και τις οικονομικές προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας για τον Μπα Σάικοτ. Μίλησες για τη βιομάζα και δεν το ανέφερα αυτό προηγουμένως, συγγνώμη. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι εν εξελίξη. Πράγματι εμείς συμμετέχουμε ιδιαίτερα στις συζητήσεις που έχουν να κάνουν με τη βιομάζα. Και αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πετύχουμε το μεγαλύτερο αντίκτυπο για τα κριτήρια αυτά βιωσιμότητας για τη βιομάζα και μέχρι τώρα η βιομάζα έχει μηδενικό βάρος στο σύστημα εκμπορίας εκπομπών. Πώς θα το συνδέσουμε αυτό με τα πολιτικά κριτήρια για τη βιομάζα. Η δική μου εντύπωση είναι όπως κάναμε και με τα βιοκάρσιμα στην Ιρλανδία. Πρέπει να πετύχουμε σωστά την πολιτική που θα κάνουμε. Είναι ενοχλητικό να έχουμε μια νομοθεσία και μια μεθοδολογία να πρέπει να την αλλάζουμε συνέχεια. Αλλά αυτός είναι κατά ανάγκη ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσουμε σε τομείς όπου ανανεώνεται συνέχεια η επιστημονική γνώση. Και πρέπει να αντανακλά την επιστημονική γνώση η πολιτική μας. Οι υπηρεσίες μας παρακολουθούν από πολύ κοντά όλα αυτά τα θέματα και είναι ιδιαίτερα ενεργές στις εσωτερικές συζητήσεις. Επίσης αυτά που είπατε για το τομέα της χαλιβουργίας. Κάναμε σαφές ότι κάποιοι τομείς που είναι ενεργοβόροι και που φοβούνται το θέμα της ανταγωνιστικότητας χάρη στην ε, άσκηση αυτή βαθμονόμησης, το benchmarking, υπήρξαν πολύ περισσότερα δωρεάν πιστοποιητικά για ορισμένου τομεί από ό,τι χρειάζονται. Είναι απαραίτητο λοιπόν εδώ πέρα να διορθώσουμε την κατάσταση. Και υπάρχουν και εσωτερικές συζητήσεις για τη χαλιβουργία. Το κύριο πρόβλημα του τομέα χαλιβουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λάθος να πούμε ότι προέρχεται από προβλήματα όπως αυτά του ETS. Είναι η υπερβολική παραγωγική ικανότητα. Είχαμε κάποια στοιχεία την προηγούμενη εβδομάδα όπου ήταν φανερό ότι οι εξαγωγές χάλιβα πήγανε μια χαρά πέρσι και κατάφεραν να υπερκεράσουν και την αύξηση των εισαγωγών. Αλλά όταν συζητάμε όλες αυτές τις κατατομίες Πολιτικέ, Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονό ότι το ενεργειακό κόστο είναι ένα βασικό θέμα και το είδαμε αυτό και στι ΗΠΑ, να απαραίτητο να το συζητήσουμε επί τη βάση πραγματικών στοιχείων και όχι επί τη βάση παραπληροφόρηση. Προσπαθούμε να το πούμε αυτό όταν έχουμε την ευκαιρία να το αναφέρουμε σε διάφορα βιομηχανικά φόρμα, αλλά είναι απαραίτητο και εσεί να έχετε επίγνωση αυτού του θέματο. Η όλη αυτή άσκηση στην οποία αποδίονται οι υπηρεσίε υπηρεσίες σε σχέση <clears throat> με τις κρατικές επιδοτήσεις για το περιβάλλον και την ενέργεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ασχολούνται ιδιαίτερα και δεν περιμένουν απλώς παθητικά δουν τι θα προκύψει. Αυτά που είπε η κυρία Χιούμπνερ, γιατί δεν αποσύρουμε την πρόταση της Κομισιόν. Καταρχήν, με κάθε σεβασμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από δύο θεσμικά όργανα που πρέπει να νομοθετήσουν επί τη βάση της πρότασής μας και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θέλει το Συμβούλιο. Αυτό είναι ένας λόγος. Επίσης, όπως είπε και ο Πρόεδρός σας, υπάρχει μια αίτηση για μια νέα, πρώτα, για μια νέα ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Το αν θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο ή α, θα το στείλει πίσω στην Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος, αυτό δεν το ξέρουμε. Γιατί λοιπόν αποσύρουμε την πρότασή μας εμείς προτείνουμε προτάσεις γιατί θεωρούμε ότι είναι πάντα η σωστή πολιτική και χρειαζόμαστε και την συμβολή των άλλων οργάνων για να δούμε κατά πόσον ευσταθούν αυτές οι πολιτικές. Τώρα για τις λεγόμενες πράσινες θέσεις εργασίας. Η κυρία Κλάσσα έθεσε και ένα ερωτηματικό δίπλα στα κριτήρια βιωσιμότητας και είπε ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται και στις εισαγωγές ώστε να μην υπάρχει κάποια διάκριση σε βάρος των ευρωπαϊκών εταιριών έναντι των ανταγωνιστών τους. <clears throat> Έχουμε αυτή τη μελέτη επίσης. που λέει η οδηγία λέει ότι βασιζόμαστε στην καλύτερη γνωσ... επιστημονική γνώση. Τώρα μπορεί κάποιοι να επιχειρηματολογήσουν με διαφορετικό τρόπο και να πούν ότι δεν θίγεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία με τον τρόπο αυτό. Και τον κύριο Γιώργενσεν, οι αντιδράσεις των άλλων εταίρων, ίσως μπορώ να σας τα πω τώρα στα δανέζικα. Να απαντήσω λοιπόν στα δανέζικα αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνουμε στον τομέα αυτό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν ήδη θεσπίσει ένα σύστημα για την εμπορία εκπομπών και είναι σαφές ότι το σύστημα αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η απάντηση και η απόφαση θα πρέπει να γίνει στο Συμβούλιο. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα ως Κομισιόν και για την αύξηση θερμοκρασίας του πλανήτη μας κατά δύο βαθμούς την προηγούμενη εβδομάδα. Υπήρξε μια μελέτη που έκανε τον κόσμο να πιστεύει ότι έχουμε περισσότερο χρόνο. Ίσως τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα από ό,τι νομίζαμε πήγα σε αυτή την επιστημονική συνδιάσκεψη στο Βερολίνο που ήταν και ο καθηγητής Χούμπερ και του τέθηκε ένα ερώτημα σε μια συνέντευξη τύπου αν μπορούμε τώρα να την αράξουμε, να χαλαρώσουμε. Και έδωσε μια πραγματική εξήγηση για το αν αυτό έχει νόημα ή όχι. Αν χίλιοι επιστήμονες μας λένε ότι αυτά τα πράγματα είναι κατεπήγοντα, ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν είναι κατεπήγον. Ήταν πάρα πολύ σαφής λοιπόν ο καθηγητής Χούμπερ είπε εξήγησε τι σημαίνουν αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε και είπε όχι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ικανότητα των θαλασσών να απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακος, αλλά αυτό είναι ένα δήμα παραπάνω της κρίσης. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας πρέπει να κάνουμε να επαναπαυόμαστε όλα αυτά λοιπόν τα οι ποσότητες του διοξιδίου του άνθρακος που απορροφούνται μας δίνουν ίσως τη δυνατότητα να πούμε ότι θα σταθεροποιηθούμε κάτω από την αύξηση, σε μια αύξηση κάτω από τους δύο βαθμούς, εάν κάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Και αν με ρωτάτε πώς εγώ απαντώ σε αυτό το ερώτημα για τους δύο βαθμούς. Μην ξεχνάτε ότι είναι μονάχα 3,5 χρόνια από τότε που οι ηγέτες του κόσμου αποφάσισαν ότι πρέπει να μείνουμε κάτω από μια αύξηση θερμοκρασίας δύο βαθμών είναι από τα λίγα πράγματα που σε επίπεδο ηγετών αποφασίστηκε για την κλιματική αλλαγή, ότι πρέπει να, μειώ, να περιορίσουμε την αύξηση θερμοκρασία σε δύο βαθμούς μονάχα Κελσίου. Τίποτα δεν έχει αλλάξει λοιπόν τη σοβαρότητα του θέματος αυτού και όταν λένε κάποιοι ότι μπορούμε απλώς ίσως να μετακινήσουμε τα τέρματα και δεν είναι τόσο σημαντικό στο στόχο των δύο βαθμών. Αυτό είναι σαν την οικονομική πολιτική. Έχουμε κάποιους στόχους, δεν τους πετυχαίνουμε, και τους μετακινούμε μετά τους στόχους μας. Όχι, πρέπει να είμαστε σοβαροί για τους στόχους που θέτουμε. Αν δεν είμαστε λοιπόν έτοιμοι να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, θα πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες. Και η τελευταία μου παρατήρηση, έχουμε το διεθνή, διεθνές πλαίσιο και το όριο των δύο βαθμών. Αλλά αν δείτε τη συνολική ανάλυση οικονομικής κατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπετε ότι υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για τους οποίους, παρά όλα αυτά που κάνουν οι ανταγωνιστές μας, ή δεν κάνουν και κάνουν πολύ περισσότερα από ό,τι εμεί πιστεύουμε μερικέ φορέ. Κάνουν πολλά πράγματα, ακόμα και αν δεν κάνουν τίποτα οι ανταγωνιστέ μα είναι προ το συμφέρον τη Ευρώπη να γίνει πιο αποδοτική σε σχέση με την ενέργεια, να εξαρτάται λιγότερα από τα ορυκτά καύσιμα και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με πολλού τρόπου. Θα ήταν ανόητο να μην το κάνουμε με έναν τρόπο ο οποίο συγχρόνω θα μα επέτρεπε να πετύχουμε του κλιματικού μα στόχου. Ευχαριστώ πολύ την κόνη Χέντεγκαρτ την Επίτροπο για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και για την ε, δέσμευση που έχει καταδείξει και την προσήλωσή της στην αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Η ανάλυση η οποία μας παρουσίασε ε, αφορά συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένες ενέργειες. Σε ό,τι αφορά την κλιματική πολιτική, βλέπουμε πολλές φορές ότι το πνεύμα ε, έχει τη θέληση αλλά η ΣΑΡΚΣ είναι ασθενής και πρέπει επομένω να φέρουμε και την σάρκα να λειτουργήσει καλύτερα και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελπίζω ότι η δική μας συμβολή θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους φιλόδοξους στόχους σας και είναι γεγονός ότι σε μια οικονομική κρίση δεν είναι πάντα εύκολο να δίνουμε την απαραίτητη έμφαση σε αυτά τα θέματα, αλλά τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε τις ε, προσπάθειες που χρειάζονται για το σύστημα εκπομπών και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, δέσμευσή σας, για την εργασία σας και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε η πρόταση για την οπισθοφόρτηση να μπορέσει να ευδοκιμήσει. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας και καλή τύχη.